Πάντοτε υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτό είναι ένα ρίσκο που είναι μέρος του σχεδιασμού ε, των δραστηριοτήτων μας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Commissioner. <clears throat> Η συζήτηση έληξε εδώ. Η επόμενη συνεδρία θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη, 19 Μαΐου από τις 9 ε, το πρωί έως τη 1 μετά τη μεσημβρία και από τις 3 έως τις 9.30 μετά μεσημβρία. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έληξη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πίτροπο, τους κυρίους και τις κυρίες συναδέλφους, τους διερμηνείς και τους συνεργάτες μας που μας συνόδεψαν μέχρι πολύ αργά. Καλή σας νύχτα.